ο κύριος είναι διαδικαστικό. Όχι, εντάξει, μετά θα πάρτε το λόγο. Στην Δευτέρα δεν έχουμε αλλαγέ για την ημερήσια διάταξη. Θα παραμείνει όσο έχει η πράσινη τώρα. Ζήτησε για να γίνει συζήτηση για τα για τη αμόλογα σταθερότητας μετά τη συζήτηση ε, για το Μαρόκο. Ζητάει κανείς από, το λόγο, από τις το λόγο. Όχι. Σωστά το είπατε. Θέλουμε επειδή είναι τρει εκθέσει και συζήτηση από την Επιτροπή Αγροτικών Ζητημάτων να συζητηθούν μαζί. Θέλουν λοιπόν οι πράσινοι να συζητηθεί το θέμα για τα ομόλογα σταθερότητα μετά τη συζήτηση για ε, το Μαρόκο, για την Ευρωπαϊκή Συμφωνία. Είναι κανείς κατά? Θέλει κανείς να πάρει το λόγο και να αντιταχθεί σε αυτή την πρόταση? Όχι. Ωραία, λοιπόν. Ποιοι είναι υπέρ της πρότασης των πρασίνων? Κατά. Αποχές. Ωραία, λοιπόν, αποφασίζεται ούτως. Θα γίνει η συζήτηση μετά την συζήτηση για την Ευρωπαϊκή, Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωση και Μαρόκο. Δεν ε, έλαβα καμία αίτηση για τροποποίηση τη ημερήσια διάταξη. Συμφωνούμε λοιπόν στην ημερήσια διάταξη ω έχει για τι υπόλοιπε ημέρε. Πολύ ωραία. Διαδικαστικό, ο κύριος Σβόμποντα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, να σας υποδείξω μια περίπτωση να σας παρακαλέσω να λάβετε τα απαραίτητα μέτρα. Κοιτώντας το website Postal Range, το οποίο υπό κανονικές συνθήκες δίνει πληροφορίες αξιόπιστες, ο Γκρους ε, δημοσιογράφος Old Bayer, έκανε κάποιες επιθέσεις κατά της Νέλης Κρούς και μάλιστα παράλογες επιθέσεις κατά των συναδέλφων ε, Λούνατσεκ. Πρόκειται για δημοσιογράφο, φυσικά μπορούμε να πούμε, αλλά πρόκειται για δημοσιογράφο, ο οποίος σύντομα, πριν από πρόσφατα μάλλον, διοργάνωσε μία διαδήλωση υπέρ του Ορμπάν, μία διαδήλωση που σύμφωνα με πολλές πληροφορίες ε, ε, εγέρθηκαν και μηνύματα αντισημητικά να ζητήσω από τον Πρόεδρο να προασπίσει την τιμή του Κοινοβουλίου και της κυρίας ε, Λούνατσεφ να ελέγξουμε αν οι μεταφράσεις που λάβαμε είναι σωστές γιατί στην περίπτωση αυτή νομίζω ότι θα πρέπει το Κοινοβούλιο μας να προασπιστεί ε, την τιμή της κυρίας Λούνατσεφ ανεξάρτητα από το ότι είμαστε υπέρ ή κατά του Ορμπάνου. Πρόκειται για παράδεκτα πράγματα. Τώρα στις επιθέσεις ε, κατά της κυρίας Νέιλι Κρούς σε ό,τι αφορά την εκπλήρωση των νόμιμων κατοικόντων της, νομίζω ότι και αυτό είναι παράδεκτο. Νομίζω ότι στην πολιτική αυτή αντιπαράθεση πρέπει να υπάρχουν κάποια φιλελεύθερα πρότυπα. Υπάρχει ένας τρόπος αντιπαράθεσης. Δεν είναι αποδεκτά πράγματα αυτό. Ο τρόπος κατά τον οποίο προβάλλεται στην δημοσιότητα στην Ουγγαρία η συνάδελφος Λούνεσεκ είναι απαράδεκτος. Ελπίζω, Πρόεδρε, να τα ερευνήσετε αυτά και αν χρειαστεί να προσπίσετε την τιμή και του Κοινοβουλίου και της κυρίας Λούνατζεκ. Ευχαριστώ κύριε Σβόμπουτα, και εννοείται ότι θα εξετάσω θα ζητήσω να μου δώσουν τα σχετικά έγγραφα και σε περίπτωση που ε, πλήττεται η τιμή και η ακαιρεότητα της κυρίας Λούνασεκ και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα λάβουμε τα απαραίτητα μέτρα για να την υπερασπίσουμε. Θα, λάβω, θα αναλάβω επαφές, ε, θα έρθω σε επαφή με τον κύριο Μπαρόσο για να δούμε μήπως πρέπει να ληφθούν μέτρα για την υπεράσπιση της τιμής της κυρίας Κρούς. Ενδεχομένως να πρέπει να ληφθούν από κοινού μέτρα. Κυρίες και κύριοι, θα ήθελα να σας αναφέρω μία περίπτωση η οποία μου ανησυχεί ιδιαίτερα.